για όλους που είναι ανθρώπινο δικαίωμα, θεμελιώδες μάλιστα. Και επίσης λέει σαφώς το κείμενο ότι η σπατάλη ύδατος πρέπει να αποφεύγεται στα κράτη-μέλη. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε και καλύτερους τρόπους μέτρησης της ποιότητας ε, του ποσίμου ύδατος. Αντιμετωπίζουμε όμως προκλήσεις. Με βάση κάποιες εκτιμήσεις το 40% του ύδατος ε, χάνεται λόγω διαρροών ε, από το σύστημα διανομής. Αυτό είναι μη βιώσιμο για το περιβάλλον και οικονομικά και για τους πολίτες μας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πολύ αυστηρότερος ε, έλεγχος και μέτρα ούτως ώστε να γνωρίζουν και οι πολίτες πόσο νερό και ποσοστό του νερού για το οποίο πληρώνουν χάνεται από διαρροές. Και επίσης χρειάζονται αυστηρότερα κριτήρια για ορισμένες ε, βλαβερές ε, ουσίες όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και επίσης πρέπει να δούμε τη συνδυασμένη δράση κάποιων χημικών. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολλή πίεση επί των ε, υδροφόρων οριζόντων από όπου παίρνουμε το πόσιμο είδωρ. Οπότε είναι η τελευταία μας ευκαιρία να δράξουμε το θέμα αυτό για να υπάρξει μια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να εγγυηθεί καθαρό πόσμο νερό, αποτελεσματική διαχείρισή του και διανομή του και είναι δική μας ευρωπαϊκή ευθύνη να φροντίσουμε να αντιμετωπιστούν ε, και οι υπάρχοντες κίνδυνοι αλλά και οι μελλοντικοί κίνδυνοι στο σύστημα διανομής. Και αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκό και όχι ε, κρατών μέλων. Χάνσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο πόσιμο είδωρ, ε, θα επιτύχουμε παράλληλα να μην πίνουν εμφιαλωμένο νερό και έτσι θα έχουμε μείωση των πλαστικών. Αυτό θα είναι καλό για το περιβάλλον και παράλληλα θα ε, εξοικονομήσουν και τα νοικοκυριά. Εάν πίνουν περισσότερο νερό από τη βρύση, θα μειωθεί λοιπόν και χρήση πλαστικών μπουκαλιών και μπορεί να εξοικονομήσουν μέχρι και 600 εκατομμύρια το χρόνο τα νοικοκυριά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι οριακές τιμές για το ε, μόλιβδο, κάποια βακτηρίδια, και του ενδοκρινικού διαταράκτε να μειωθούν για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι συμπολίτε μα στην ποιότητα του νερού. Το πλαστικό στο νερό είναι ένα πρόβλημα τόσο σημαντικό και αυξανόμενα σημαντικό. Γι' αυτό κυρίω πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα μικροπλαστικά, το οποίο πρόβλημα δεν έχει γίνει αντικείμενο επαρκού έρευνα, αλλά μπορεί να έχει σοβαρέ επιπτώσει και είναι λυπηρό που τα κράτη-μέλη δεν κατέληξαν ε, συντομότερα σε μια κοινή στάση. Και επέτρεψαν περιορισμένες απαιτήσει για την πρόσβαση στο νερό. Θα ήταν σημαντικό εν ώψη και της Παγκόσμιας Μέρας Ήδατος στις 22 Μαρτίου να είχαμε ολοκληρώσει την εξέταση αυτής τη οδηγία. Αλλά δεν είναι δική μας ευθύνη. Και ευχαριστώ τον συνάδελφο Μισελ Νταντά και τους συνεργάτες του για την καταπληκτική εργασία, αλλά λυπάμαι για αυτούς που θα καταψηφίσουν την έκθεση γιατί είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Σόιντροβα. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, δικαιοκριμένοι συνάδελφοι. Το νερό είναι ζωή. Είναι ένα στατηγικό υλικό, στατηγικό αγαθό και πρέπει να το προσέχουμε καλύτερα. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης υπάρχουν χώρες και περιοχές όπου το πόσιμο νερό σπανίζει και θα πρέπει να εισάγεται από πιο απομάκρες περιοχές. Το νερό γίνεται ε, μια πρώτη ύλη στρατηγικής σημασίας. Καλωσορίζω συνεπώς την Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία ε, αναβαθμίζει και αλλάζει την προσέγγισή μας όσον αφορά το νερό μετά από 20 χρόνια. Υποστηρίζω και τους τέσσερις τομείς δράσης την αξιολόγηση βάση κινδύνου, βελτίωση της διαφάνειας, πρόσβαση στις πληροφορίες και η ποιότητα επίσης των υδάτων και των υλικών. Χρειάζεται, χρειάζονται αυστηρότερες προδιαγραφές όσον αφορά διάφορους συντελεστέ, διάφορες ουσίες. Είναι κάτι σημαντικό. Αλλά δεν θα πρέπει να αυξηθεί το τίμημα που πρέπει να καταβάλλεται για το νερό. Όμως η ανθρώπινη υγεία είναι η βασική μας ε, βασικό μας μέλημα και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Βέβαια, τα κράτη-μέλη από παραμένουν υπεύθυνα για την ποιότητα των υδάτων, άρα εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης και όσον αφορά την πρόσβαση στο νερό. Χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται επαρκής ενημέρωση προς τους ε, καταναλωτές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει επίσης να είμαστε και οικονόμοι όσον αφορά το νερό. Και χάρη στα διαθωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μεταξύ άλλων, πολλά κράτη-μέλη έχουν βελτιώσει ε, την ε, κατεργασία των ε, υδατίνων λιμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε το νερό για την υγεία όλων μας. Συνάδελφε Ρούμπη, για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας, ε, κύριο Νταντά, ιδιαίτερος. Το νερό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής επιβίωσής μας. Και κυρίως μας ενδιαφέρει το πόσιμο είδωρο. Και χαίρομαι, χαίρομαι που στις 3 Απριλίου, στις 4.30 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, την επόμενη εβδομάδα, θα παρουσιάσουμε την έκθεση των ΟΕΕ για το νερό. Νομίζω ότι θα είναι μια ιστορική στιγμή και από πλευράς πολιτικής ανάπτυξης τονίζω ότι οι βιώσιμοι στόχοι ανάπτυξης έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όλοι γνωρίζουμε. Χωρίς νερό δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη διατροφή. Η παραγωγή τροφίμων χρειάζεται νερό. Και αν δεν έχουμε επαρκή τρόφιμα δεν θα επιτύχουμε και το στόχο 7 για τις βιώσιμες ε, ενέργειες. Γι' αυτό οι στόχοι 5, 6 και 7 είναι αλληλοσυνδεδεμένοι και έτσι θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, όπου χρειάζονται αυτές οι υποδομές. Σήμερα 50% το πληθυσμού μας ε, χρειάζεται να αγοράσει νερό λόγω της κακής ποιότητας ε, του νερού της βρύσης του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ε, μια συνέχιση της πολιτικής μας προς αυτή την κατεύθυνση και να βοηθήσουμε και τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ξέρετε ότι εκατομμύρια ανθρώπων δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια νέα προσέγγιση για να επιτύχουμε τον ε, στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης 6, να έχουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να επενδύσουμε παγκόσμια για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ε, έχουν καλύτερη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Σας ευχαριστώ για τη διαδικασία. Κάτσε τη Άι, Συνάδελφε Φαρία, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Νταντά για το εξαιρετικό του έργο. Ε, υπενθυμίσω και εγώ την πρωτοβουλία πολιτών Right Water. Ήμουν αισιόδηση εισηγητής ε, για αυτήν και αυτό που έλεγε είναι ότι μέχρι το 2030 πρέπει να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο 6 από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλουμε η ποιότητα των υδάτων, είναι κάτι το οποίο να μπορούμε να εγγυθούμε στους πολίτες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και πρέπει να αποφύγουμε να μην υπάρχει αρκετό πόσιμο νερό. Κάτι το οποίο θα αποτελέσει όμως πρόκληση για μας και δυσκολία δεδομένων των κλιματικών αλλαγών. Εμείς πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ποιότητα του ύδατος και για την ε, πρόσβαση που προσφέρουμε στο είδωρ. Οι πολίτες που είναι καταναλωτές ε, πρέπει να καταλαβαίνουν ότι προστατεύονται τα δικαιώματά τους στην πρόσβαση σε νερό ποιότητας. Πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε το νερό αυτό. Είναι θέμα δημόσιας υγείας αλλά και δικαιοσύνης, κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα την παρέμβαση του Επιτρόπου του κυρίου Αβραμόπουλου. Κύριε Αβραμόπουλο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που άκουσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επιβεβαιώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει προς το συμφέρον των πολιτών μας και ότι όλοι στηρίζουν τον στόχο αριθμό 6 βιώσιμης ανάπτυξης που αναφέρεται στην πρόσβαση στο νερό. Ελπίζω όλα αυτά να αντικατοπτριστούν και στην πρώτη ανάγνωση, ώστε να αρχίσει ο τριμερής διάλογος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με φιλόδοξες θέσεις σε σχέση με την ποιότητα των υδάτων, την προστασία της υγείας και την πρόσβαση στο νερό. Επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει τους συνομοθέτες προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία η οποία να στηρίζει τους στόχους που είναι κοινοί μεταξύ μας και θα φροντίσουμε έτσι οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους την υψηλότερη δυνατόν ε, ποιότητα και προστασία τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και για την δέσμευσή σας υπέρ του σκοπού αυτού. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα θα ακούσουμε την παρέμβαση του εισηγητού του κυρίου Νταντέν. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, πράγματι είναι η τελευταία φορά που παρουσιάζω μία έκθεση εδώ στο σώμα. Και έτσι θέλω να σας πω ότι έχω μέσα μου μετά από διάφορες μισές αλήθειες που ακούσαμε σήμερα. Όταν μιλάμε για την τιμή του νερού, δεν μιλάμε για την τιμή του νερού. Μιλάμε για την τιμή των σωλήνων, των κέντρων ίδρευσης, της διανομής, του ελέγχου των αναλύσεων. Και εντάξει, ναι, δύο εκατομμύρια περίπου πολίτες υπέγραψαν πράγματι την πρωτοβουλία για να έχουν όλοι πρόσβαση στο νερό. Και όλοι συμφωνούμε με το στόχο αυτό. Όμως, ακούω και τα εκατομμύρια πολίτες που μας ζητούν να είναι φτηνό το νερό. Δηλαδή, να υπάρχουν οι καλές υποδομές για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, ο καταναλωτής και να προστατεύεται η υγεία του. Οπότε, πώς θα γίνει. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Τα έχουμε αυτά τα δεδομένα και συμπεριλαμβάνονται στα ευρωπαϊκά κείμενα. Και όταν ε, ακούμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορες παραμέτρους, ναι, αλλά ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα πρέπει να μας προτείνει μία μέθοδο έγκρισης που να συνάδει με την ανθρώπινη υγεία. Και για τα μικροπλαστικά δεν έχουμε αυτή τη μέθοδο αξιολόγησης, ούτε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες δεν έχουμε αυτή τη μεθοδολογία. Ναι, φυσικά και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα, γιατί το νερό είναι αναγκαίο για τη ζωή και γιατί η πρόσβαση σε νερό ποιότητας για όλους όντως πρέπει να είναι μια απέτηση. Αν καταφέρουμε λοιπόν να βελτιώσουμε το νερό της βρύσης και αν πείσουμε τους πολίτες ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θα έχουν πρόσβαση σε νερό ποιότητας, τότε ναι, θα καταργηθούν τα πλαστικά μπουκάλια. Και βέβαια ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι το νερό της βρύσης τους ε, κοστίζει πολύ λιγότερο από ότι το νερό που αγοράζουν ε, σε μπουκάλια ε, τα οποία εμπιστεύονται απόλυτα παρόλο που εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είσαστε η μόνη εδώ στο σώμα που έχετε μπροστά σας ένα ποτήρι νερό. Ε, λοιπόν, σηκώστε αυτό το νερό στην υγεία όλων αυτών των εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για νερό ποιότητα. Εγώ εμπιστεύομαι αυτού που θα μα διαδεχθούν εδώ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Τώρα, πέρα τούτη η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την κοινή συζήτηση όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των σημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έκθεση μέλο και Λέναρτς. Το λόγο έχει ο συγητής Λέναρτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, με την νομοθεσία αυτή κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να είναι περισσότερο ασφαλής η Ευρώπη ώστε να αποφεύγουμε τους εγκληματίες και τους δρομοκράτες, να μπορούμε πιο γρήγορα να τους συλλαμβάνουμε είναι πιο αποτελεσματικές οι μέθοδοι ελέγχων, προστατεύουμε καλύτερα τα σύνορά μας, ε, εντοπίζουμε ψεύτικες ταυτότητες. Εδώ στο Στρασβούργο, λίγα χιλιόμετρα από αυτόν εδώ το χώρο, εκεί όπου βρίσκεται η έδρα της Λίζα, εκεί ο κόσμος ασχολείται με την ασφάλεια, την ασφάλειά μας. Οι προδιαγραφές είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Όμως δεν υπάρχει τρόπος ο οργανισμός αυτός να επικοινωνεί με άλλους αντίστοιχους εθνικούς στην Ευρώπη ή με άλλους που ασχολούνται με την ασφαλειά μας. Και αυτή είναι η αδυναμία του συστήματός μας μέχρι τώρα, την οποία διορθώνουμε με την πρότασή μας αυτή. Μπορούμε η, να φροντίσουμε η αστυνομία, τα τελωνία, πατώντα ένα κουμπί να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ό,τι πληροφορίες χρειάζονται και να ζητάνε και τις σωστές πληροφορίες για αυτό που χρειάζονται για να μπορούν να κάνουν καλά την δουλειά τους. Είτε πρόκειται για τα βιομετρικά στοιχεία, είτε πρόκειται για την αναγνώριση ταυτότητας, προσώπου, με ένα κουμπί μπορούν όλα αυτά τα στοιχεία να τα έχουν στη διάθεσή τους και θα είναι περισσότερο φτηνό το σύστημα και περισσότερο ασφαλές. Δεν θα χρειάζεται κάθε φορά ξανά και ξανά να ε, επανεφεύρουμε τον τροχό. Είναι περιττό όπλός να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά εργαλεία. Έπειτα, για να, αποφεύγετε ή να αποφεύγουμε τις πολλαπλές ε, ταυτότητες, θα έχουμε τα βιομετρικά στοιχεία και θα μπορούμε έτσι να ελέγχουμε αυτούς που έρχονται στην Ευρώπη με την πρόταση αυτή μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε τη δουλειά μας, μπορούμε πιο εύκολα να ελέγξουμε τα δεδομένα, μπορούμε πιο εύκολα να ελέγχουμε την πρόσβαση σε πληροφορίες και πιο εύκολα να ελέγχουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν ε, ε, χαρτιά να παρουσιάσουν στο δρόμο, αλλά εμείς μπορούμε να εντοπίσουμε την ταυτότητά τους. Είδαμε ότι οι εγκληματίες μπορούν πολύ εύκολα να φτάσουν να έχουν 20 διαφορετικές ταυτότητες στη διάθεσή τους. Ε, αυτό τώρα δεν θα μπορούν πια. Τρομοκράτες με 14 διαφορετικές ταυτότητες ε, κυκλοφορούσαν. Τώρα με αυτά τα καινούργια εργαλεία μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε. Με μια τέτοια πρόταση μόνο μπορούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχαμε μέχρι τώρα. Η ασφάλεια πηγαίνει βέβαια χέρι-χέρι με την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Και τι κάναμε λοιπόν, φροντίζουμε ναι, να έχουμε περισσότερα δεδομένα, να συγκεντρώνουμε περισσότερα δεδομένα, αλλά να τα χρησιμοποιούμε και καλύτερα. Να υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές για το πώς χειριζόμαστε το σύστημα. Και έχουμε νέα νομοθεσία που επιτρέπει στους πολίτες να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους. Αυτή η πρόταση, αυτή η νέα πρόταση είναι ένα νέο πνεύμα, ένα νέο τρόπος εργασίας που θα μας βοηθήσει τα επόμενα χρόνια και θα αποφέρει σίγουρα καρπούς. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αβραμόπουλο για την ε, εργασία του σε αυτό το φάκελο και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μέλο αλλά και όλους τους συναδέρφους και συνεργάτες μας και συμβούλους μας που όλο αυτό το καιρό μας βοήθησαν να, να καταλήξουμε σε μια καλή πρόταση. Αυτή η διαλειτουργικότητα είναι κάτι το οποίο θα μας προσφέρει μια ασφαλή Ευρώπη για να προστατεύουμε τους πολίτες μας, την αστυνομία στους δρόμους, τα τελωνία, όλοι θα συνεισφέρουν για την ασφάλεια αυτή και θα έχουν στη διάθεσή τους τα σωστά εργαλεία για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον άλλο εισηγητή, στον κύριο Μέλο. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, περί τίνος πρόκειται. Είναι η πρόσβαση στην ε, πληροφορία. Σε πολύ σημαντικέ μάλιστα πληροφορίε, τι κατάλληλε και που πρέπει να γίνεται γρήγορα και συστηματικά και αποτελεσματικά, αλλά με ελεγχόμενο τρόπο, με του σωστού ελέγχου. Όλα αυτά είναι ουσιώδη για να ελέγχουμε τα εξωτερικά μα σύνορα, για να καταπολεμάμε την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία. Σήμερα είναι ακόμη πολύ δύσκολο να ανοιχνεύσουμε, για παράδειγμα, ορισμένε περιπτώσει πολλαπλών ταυτοτήτων, δηλαδή ατόμων που έχουν πολλέ ταυτότητε. Ή διάφορε άλλε παρανομίε ε, που διαπράττονται με διαφορετικέ ταυτότητε. Ε, ε, ορισμένα στοιχεία τα έχουμε στο ΣΥΣ και στο ΕΤΙΑΣ. Δεν δεν υπάρχει πληροφορία. Το θέμα που τίθεται είναι το ότι δεν ε, την, ε, τις μοιράζονται όλοι αυτές τις πληροφορίες. Ο καθένας περιχαρακώνει τις πληροφορίες που έχει στο δικό του σύστημα, στο δικό του φορέα, ε, στο δικό του επάγγελμα, τον δικό του επαγγελματικό χώρο. Οι διάφοροι φορείς δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες γιατί δεν τους υποχρεώνει κανείς. Ενώ υπάρχουν τρόποι. Γι' αυτόν τον τρόπο λοιπόν εργαστήκαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ ως Κοινοβούλιο και με τρόπο απόλυτα ανοιχτό, ειλικρινή. Ο καθένας ε, συνέβαλε και, και ο συνεισηγητής μου, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, και οι Σκιώδης. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Κίν και τον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Και οι δύο συμμετείχατε στη συνεδριά μας και δώσατε αποφασιστικές απαντήσεις, ιδιαίτερα από πλευράς διοργανικής. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν απέδειξαν ότι όταν ε, καθορίζουμε σαφώ τι προτεραιότητέ μα, μπορούμε να δώσουμε τι καλύτερε δυνατέ απαντήσει προ το συμφέρον των ε, συμπολιτών μα. Και αυτό έγινε και εδώ. Είναι πολύ τεχνική αυτή η έκθεση, υπερβολικά θα έλεγα τεχνική, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να μάθουμε τα περίπλοκα αυτά θέματα, τα εξετάσαμε συγκεκριμένα και πιστεύω ειλικρινά ότι όταν θα εφαρμοστούν αυτά που αποφασίζουμε, οι συμπολίτε μα θα είναι σε καθεστώ μεγαλύτερη ασφάλεια. Για παράδειγμα, αυτέ οι πολλαπλέ ταυτότητε σε μία από τι τρομοκρατικέ επιθέσει στην Γερμανία, ένα από του τρομοκράτε είχε ζητήσει άσυλο. Με 14 διαφορετικέ ταυτότητε. 14. Και σε μια άλλη περίπτωση στη Γαλλία, ένα από του τρομοκράτε, την Ίσιο, είχε ε, καταγραφεί ε, σε διάφορε βάσει δεδομένων με 7 διαφορετικέ ταυτότητε. Ε, εντυπωσιακά δεν αυτά τα στοιχεία. Τέτοιε περιπτώσει ε, δεν καταλαβαίνουν οι συμπολίτε μα. Πώ μπορεί να συμβαίνουν. πώ είναι δυνατόν να γίνεται μια τρομοκρατική επίθεση στην Γαλλία ενώ υπήρχαν προφορίες για τα άτομα που την διέπραξαν στο Βέλγιο αλλά δεν είχε περάσει αυτή η προφορία στη Γαλλία. Δεν είχε γίνει ανταλλαγή προφοριών. Και δεν είναι επειδή δεν υπάρχει καλή βούληση, αλλά γιατί δεν υπάρχουν τα συστήματα, τα γρήγορα αποτελεσματικά συστήματα που να επιτρέπουν οι αρχές να λαμβάνουν ε, σε συνθήκες νομιμότητας και με προστασία των δεδομένων να λαμβάνουν τα στοιχεία. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να ελέγχουμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας, να καταπολύσουμε την κλιματικότητα, την τρομοκρατία. Όλα αυτά πρέπει να είναι πρωταρχική προτεραιότητα. Γιατί αν δεν είναι προτεραιότητα, η απουσία απάντηση από πλευρά μας, δυστυχώ αργότερα θα μετατραπεί σε θύματα σε αδικήματα που δεν πραχθούν. Εμείς εκλεγήκαμε ούτως ώστε όσο μπορούμε να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτή τη μάχη. Και είμαι πολύ περήφανος που ολοκληρώνεται αυτή η θητεία, εγώ ολοκληρώνω αυτή τη θητεία ως συνεισηγητής για αυτή την πρωτοβουλία και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό, ενώ υπήρχαν πολλές αμφιβολίες στην αρχή. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ το λόγο στον Επίτροπο τον κύριο Βραμόπουλο και μετά στον Επίτροπο τον κύριο Κίνγκ που τον ευχαριστώ για την εδώ παρουσία του απόψε. Έχετε το λόγο κύριε Βραμόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για τη φιλοξενία. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομβική στιγμή. Πιθανότατα, διότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αναμένει. Την περασμένη φορά που μάλλον είναι η τελευταία φορά που συζητούμε αυτή την πρωτοβουλία την ασφάλεια στην Ολομέλεια και είναι μια ευκαιρία να προβληματιστούμε κατανοώντας πόσο έχουμε προχωρήσει την τελευταία πενταετία. Από την αρχή που συζητήσαμε στην Ολομέλεια το θέμα, προς το τέλος του 2014, είδαμε ότι υπήρχε πράγματι ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται τα κράτη-μέλη για θέματα ασφαλείας για να ξεπεράσουμε τα διάφορα ταμπού ε, όσον αφορά την ασφάλεια του παρελθόντος και να εξετάσουμε τα θέματα εσωτερικής ασφαλείας συλλογικά, σαν ευρωπαϊκό θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ε, συνεχώς στενότερη συνεργασία. Εν αυτή τη ενία η σημερινή συζήτηση είναι έξοχο παράδειγμα της πρόοδου που έχει επιτευχθεί αυτή την πενταετία. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μας πληροφορικής για τα σύνορα, για τη μετανάστευση και για την ασφάλεια είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Η διαλειτουργικότητα είναι μία άσκηση στο να καταργηθούν τα στεγανά. Για, είναι ένα θέμα που είναι τεχνικής φύσεως, αλλά είναι η αλλαγή που χρειαζόμαστε για να αυξήσουμε την ασφάλεια της πολίτες στην Ευρώπη, για να προστατεύσουμε και διαχειριστούμε καλύτερα τα κοινά μας εξωτερικά σύνορα και να διαχειριστούμε καλύτερα τη μετανάστευση. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τους συνεισηγητές, τον κύριο Λένερς και τον κύριο Μέλο, καθώς και προς όλους τους κοιόδης εισηγητές και τους βοηθούς αυτών, διότι κατανόησαν τη σημασία της προτάσεως που υποβάλαμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο περίπου. Η διαλειτουργικότητα είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την καταπολέμηση του κατακαιρματισμού των προσπαθειών. Να κλείσουμε τα κενά της ενημέρωσης των πληροφοριών και να αντιμετωπίσουμε ε, το πρόβλημα της διαλέψεως τρομοκρατών και εγκληματιών από τα σύνορα των, ε, της Ευρωπαϊκής Αυτή είναι η καλύτερη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην καλύτερη της επίδοση. Βοηθούμε τους αστυνομικούς μας, τους μεθοριοφύλακες, τους δίνουμε τα κατάλληλα εργαλεία να κάνουν τη δουλειά τους, να μπορέσουν να προστατεύσουν τους πολίτες. Η διαλειτουργικότητα δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αποφασιστικό βήμα για αποτελεσματική πραγματική ένωση ασφαλείας διαχειριζόμενοι τα προβλήματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης με έναν ολιστικό τρόπο. Όλα αυτά εξασφαλίζοντας παράλληλα κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας με την μεγάλη σας συνεισφορά ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα γίνονται πλήρως σεβαστά. Η διαλειτουργικότητα δεν είναι ο μεγάλος αδελφός ούτε είναι μια τεράστια βάση δεδομένων και τίποτα δεν αλλάζει όσον αφορά την πρόσβαση κάθε αρχής, κάθε αξιωματούχου στα διάφορα στοιχεία που έχουμε στα συστήματά μας της πληροφορικής. Η Υπηρεσία Θεμελιών Δικαιωμάτων συμμετέχει και η Υποπτική Αρχή για τα Προστασία των Δεδομένων συμμετείχαν στην προετοιμασία της πρότασής μας. Αυτό έδειξε λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι ασφάλεια και ιδιωτικότητα είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δύο μπορούν και πρέπει να εξασφαλίζονται. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι πολίτες μας επιθυμούν περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερη Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια. Το βλέπουμε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση. Το ακούμε κάθε φορά που συναντούμε τους πολίτες μας. Η διαλειτουργικότητα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο χρήσεως των πληροφοριών για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για να πετύχουμε την ασφάλεια των πολιτών. Σε μια εκλογική χρονιά αυτό δεν θα μπορούσε να είναι κάτι πιο σημαντικό. Ε, ασκούμε πραγματική δράση, κάνουμε κάτι ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες των πολιτών μας. Όλοι μπορούμε και σωστά υπερήφανοι για αυτό το επίτευγμα. Ευχαριστώ ειλικρινά όλους αυτούς που συνέβαλαν τους δύο έξοχους συνεισηγητές, τον κύριο Μέλο και τον κύριο Λέναρς και βέβαια ευχαριστώ τον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Τζούλιαν Κίνγκ για την αφοσίωσή του, την προσπάθεια που έκανε, την αποφασιστικότητα που έδειξε για να ηγηθεί των προσπαθειών που καταβάλαμε για να καταλήξουμε στο έξοχο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Αβραμόπουλε, κύριε Επίτροπε. Και τώρα Επίτροπο ο κύριο Κίνγκ. Έχετε το λόγο. Ορίστε κύριε Κίνγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, με ευρωβουλευτέ. Θα μπορούσαμε να είχαμε βρει ένα καλύτερο όνομα. Η διαλειτουργικότητα όμως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για τους λόγους που ακούσαμε αρχίσαμε να ρωτάμε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, τι χρειάζονται. Και εκείνοι απάντησαν ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά το χειρισμό, την χρήση των πληροφοριών. Και υπήρχε μια δυσκολία στον εντοπισμό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν πολλαπλές ταυτότητες. Και ακούσαμε ότι είναι κάτι το οποίο οδήγησε σε τρομοκρατικές ε, επιθέσεις, δυστυχώς. Ένας από τους λόγους για τους οποίους νιώθουν απογοήτευση αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή είναι ακριβώς γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν τις διάφορες βάσεις δεδομένων της Ευρώπης, είτε πρόκειται για την ασφάλεια είτε για οτιδήποτε, ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα ή δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα με τον τρόπο που θα τους εξυπηρετούσε για τις ανάγκες τους. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα κάνουμε κάποια βήματα για να τους βοηθήσουμε, να κάνουν τη δουλειά τους καλά και έτσι να μας προστατεύουν, είτε πρόκειται για του συνοριοφύλακε, είτε για άλλου να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα τις πληροφορίες που διαθέτουμε στα συστήματά μα. Να βρούμε τρόπου, δηλαδή να καλύψουμε τα κενά, τι ε, τρύπε, ό,τι έλειπε. Αυτό λοιπόν τώρα περιμένουν και οι πολίτες από εμά όπως υπογράμμισε και ο κύριος Αβραμόπουλος. Νομίζω ότι πολλοί πιστεύουν ότι ήδη το κάνουμε, ήδη μπορούμε να το κάνουμε, ότι υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κάνουμε τα βήματα που χρειάζονται ακόμα. Ευθύ εξ αρχής πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλά περίπλοκα και ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε για να πετύχει αυτή η πρόταση. Και ακριβώς αυτό νομίζω ότι κάνει πρόταση και το αναγνωρίζουμε όπως το και όσοι πήραν το λόγο πριν ότι τα καταφέραμε συνεργαζόμενοι ικανοποιητικά μεταξύ μας. Η ΛΥΜΠΕ, όλοι οι ευρωβουλευτέ, το Συμβούλιο, ε, ο επόπτης ε, προσωπικών δεδομένων, όλοι από την πρώτη μέρα συνεργαστήκαμε μεταξύ μας. Για μένα αυτό είναι κάτι ακόμα θετικό, γιατί δείχνουμε ότι μπορούμε να ενσωματώσουμε όλες αυτές τις διαφορές που υπάρχουν ήδη από την αρχή και να λάβουμε υπόψη μας όλες τις θέσεις και τις ανησυχίες των διαφόρων κλάδων και να συγκεράσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως λέει ο επόπτης προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια, όλα. Και έτσι έχουμε την ευκαιρία να ελέγχουμε ότι η δουλειά που γίνεται σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό που πετύχαμε μαζί θα βελτιώσει την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων Σέγγεν και θα ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια σε όλες τις χώρες μας. Οι συναριοφύλακες, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση του νόμου, θα έχουν εύκολα πρόσβαση στην πληροφορία που διαθέτουμε και την οποία έχουν δικαίωμα να βλέπουν και όταν κάποιος ε, καταγράφεται με πολλαπλές ταυτότητες αμέσως θα εντοπίζεται. Διευκολύνεται επίσης ε, τα ταξίδια ε, για τους καλόπιστους πολίτες. Διασφαλίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κάνουμε μόνο ότι είναι αναγκαίο και αναλογικό. Δεν θα συλλέγονται στοιχεία ε, για κανένα άλλο λόγο εκτός από αυτή τη διαλειτουργικότητα. Και επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι ο έλεγχος από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο φάκελο αυτό έχει διευκρινίσει πράγματα και έχει φροντίσει για δικλείδες ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην πληροφορία. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Το αποτέλεσμα πάντως είναι μια ισχυρή νομοθετική πρόταση η οποία διασφαλίζει την προστασία στις χώρες μέλη, χρησιμοποιεί την τεχνολογία αλλά συμπεριλαμβάνει και ρήτρες ασφαλείας για να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία, να το πω αυτό σε προσωπικό επίπεδο, με τους δύο εισηγητές, τον κύριο Λέναρτς και τον κύριο Μέλο και με τους συνεργάτες τους. Ξέρω ότι δεν ήθιστε εδώ, αλλά επιτρέψτε μου δύο δευτερόλεπτα μόνο να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δούλεψαν σκληρά. Ώρες και ώρες. Όλοι μαζί καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα και άπαξ και εγκριθεί η νομοθεσία αυτή. Από εκεί και πέρα όλοι μας πρέπει να φροντίσουμε ώστε να εφαρμοστεί και σωστά. Το Ιγιουλίσα, για παράδειγμα, που ξέρω ότι στηρίζετε εσείς, ε, θα μπορέσει να δουλέψει καλύτερα. Όλα αυτά τα μέτρα πάνω στα οποία συμφωνούμε τώρα θα τεθούν σε εφαρμογή στην πράξη. Οι καινοτομίε που προβλέψαμε και που υπογραμμίσατε κι εσείς θα κάνουν τη διαφορά όσον αφορά την ασφάλεια επιτόπου μόνο εφόσον και αν εφαρμοστούν πλήρως. Συλλογικά λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μεμονωμένα στην κάθε χώρα μέλος. Και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέλει να συνεχίσει να παρακολουθεί το πώς προχωράει το θέμα αυτό και η εφαρμογή των μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξέρετε ότι θα φροντίσει για τη στήριξη και για τη χρηματοδότηση και δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες μας ώστε οι χώρες μέλη να ε, τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν λάβει είναι καλό για την ασφάλεια όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε Κίνγκ. Και τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Σε αυτό το στάδιο δεν δεχόμαστε γαλάζιες κάρτες. Συνάδελφε Ράντεφ, για τρία λεπτά έχετε το λόγο, εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Αβραμόπουλε και κύριε Επίτροπε Κίνγκ, κυρίε και κύριοι, καταρχά ευχαριστώ του συζητητέ για την εργασία του για την έκθεση αυτή. Οι τρομοκρατικέ επιθέσει των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι υπάρχουν ανεπάρκειες στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας. Οι διάφορες αστυνομικές αρχές και οι αρχές ασφαλείας έχουν ε, πλήθος προφοριών, αλλά δεν υπάρχει ανταλλαγή τους, γιατί δεν υπάρχει ένας κατάλληλο μηχανισμός. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, εφαρμόσει διάφορα συστήματα, αλλά το καθένα έχει συγκεκριμένο λόγο λειτουργίας και ε, δεν ανταλλάσσει προφορίες. Δεν ελέγχουν δηλαδή τις άλλες υπηρεσίες αν έχουν ε, σχετικές προφορίες. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να υπάρξει αυτή η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Δηλαδή, είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε ότι οι διάφορες βάσεις δεδομένων το ΒΙΣ, το ΣΕΝΓΕΝ και άλλες βάσεις δεδομένων πρέπει να επικοινωνούν. Ούτως ώστε ένας ε, συνοριοφύλακας ή ένας αστυνομικός όταν ελέγχει ένα άτομο να μπορέσει εύκολα να διαπιστώσει εάν σε κάποια από τα συστήματα υπάρχει μια ειδοποίηση, ένα συναγερμός για αυτό το άτομο. Χαίρομαι που τώρα οι αρμόδιες αρχές θα είναι σε θέση να κάνουν ε, συνολικούς ελέγχους λοιπόν υπόπτων με βάση τα βιομετρικά του στοιχεία και όλα τα άλλα στοιχεία για το άτομο αυτό. Έτσι θα μπορέσουν να ανοιχνεύσουν πολλαπλέ ταυτότητε, για παράδειγμα και να συγκρίνουν την πληροφορία και τα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν καλύτερα εάν το άτομο αυτό είναι κίνδυνος για την ασφάλεια τη Ευρώπη. Χωρί ωστόσο να παραβιάζουν τα δικαιώματα αθώων ταξιδιωτών θα υπάρχουν όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Γιατί μόνο οι εξοδοτημένοι υπάλληλοι θα έχουν ε, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την ανταλλαγή στοιχείων. Τα κράτη-μέλη πρέπει λοιπόν να ε, εισάγουν στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Δεδομένων στοιχεία υψηλής ποιότητας και τους αναγκαίους συναγερμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ντάλι δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητάμε ε, ένα θέμα που δεν ήταν εύκολο. Ο συνάδελφος ε, από την ομάδα των σοσιαλιστών αλλά και εγώ κάναμε ό,τι μπορούσαμε ούτω ώστε οποιοδήποτε συμβασμό ο οποίο επετεύχθη να εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όχι μόνο των συμπολιτών μα, αλλά και οποιοδήποτε έχουμε συλλέξει στοιχεία. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι ένα σύστημα συλλογή πληροφοριών μεγάλη κλίμακα και ω ομάδα ποτέ δεν θελήσαμε να υποχωρήσουμε από τι αρχέ του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των συμπολιτών μα. Για μα η ασφάλεια ήταν πάντα προτεραιότητα. Αλλά είναι και η προστασία των δεδομένων επίση προτεραιότητα. Κατά τι διαπραγματεύσει, πάντα θέλαμε να διασφαλίσουμε ουσιαστική και αποτελεσματική ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των διαφόρων ε, βάσεων δεδομένων για τους αστυνομικούς, ε, τους υπεύθυνους για την ε, μετανάστευση, τους ε, προξενικούς υπαλλήλους, τους ε, συνοριοφύλακες. Γι' αυτό ως ε, σοσιαλιστική ομάδα επιμείναμε ιδιαίτερα στι στις μη διακρίσεις και την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ούτω ώστε να προστατεύουμε τον ιδιωτικό βίο των συμπολιτών μα. Γι' αυτό θέλουμε και να υπάρχει αυτή η δικτυακή πύλη που θα επιτρέπει τους πολίτες να διαπιστώνουν αν τα δεδομένα τους δεν έχουν ε, αποθηκευθεί σωστά στις τράπεζες δεδομένων. Το κάναμε αυτό ούτως ώστε οι πολίτες που θέλουν να αμφισβητήσουν ε, λανθασμένα στοιχεία να έχουν δυνατότητα να ξέρουν σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούν για να διορθωθούν τα στοιχεία τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ναι μεν προστατεύουμε την ασφάλεια χωρίς όμως να θέσουμε κατά μέρο τα δικαιώματα των πολιτών που εργάστηκαν τόσο σκληρά οι πολίτες για να τα αποκτήσουν. Και μεταξύ αυτών είναι και η προστασία των δεδομένων. Η ισορροπία μπορεί πάντα να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Στίβεν. Κυρία Στίβεν, μισή λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νομοθετικό πακέτο για την διαλειτουργικότητα, ε, για την συνδεσιμότητα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι τράπεζες δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούνται καλύτερα και στα συστήματα συνόρων και θεωρήσεων. Κάποιο απ' έξω που παίρνει μια βίζα για να έρθει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι τρομοκράτης, δεν είναι κανένας παράνομος, ότι θα μπορεί να τον παρακολουθήσουμε και να το εντοπίσουμε αυτό. Θα μπορούν λοιπόν όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα από τις αρχές μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ώστε να εντοπίζουν για ποιον πρόκειται. Όταν ε, οι αστυνομίε ε, στο εξωτερικό δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, μέσω αυτών των συστημάτων διαλειτουργικότητας θα μπορούν πια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται όλο και περισσότερους μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απειλούν μια συνεχή ε, απειλή για την ασφαλειά μας. Μέσω της σύνδεσης των συστημάτων ε, αυτών θα προστατεύεται καλύτερο ο χώρος μας. Έτσι θα προσφέρουμε καλύτερη προστασία στους πολίτες μας από την παράνομη μετανάστευση. Το κείμενο αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ταυτοτήτων και δεν πρέπει να ξεχνάμε συγχρόνως ότι η προστασία των δεδομένων είναι κάτι που επίσης διασφαλίζεται με την πρόταση αυτή. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει με μεγάλη πλειοψηφία αυτή την νομοθετική πρόταση και οι χώρες μέλη επίσης να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ, έχει το λόγο. Ζεράρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριοι Επίτροποι. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής. Για μία μόνο συζήτηση έχουμε δύο επιτρόπους που συνομιλούν, δεν ακούνε τίποτα. Τέλο πάντων, έχουμε τη χαρά του, έχουμε εδώ. Δεν θέλω να κρύψω τη χαρά μου. Αν υπάρχει ένα θέμα για το οποίο ήθελα να καταλήξουμε κάπου σε αυτή τη θητεία είναι αυτό της διαλειτουργικότητας. Λοιπόν, εξυγχρονίσαμε τα τελευταία χρόνια κάποια συστήματα, το VIS, το ACS, το Eurodac, το ETIAS και άλλα αλλά αυτά τα συστήματα δεν έχουν καμία διασύνδεση μεταξύ του, οπότε μείωσε την αποτελεσματικότητα τη χρήση των δεδομένων που συλλέγουμε και χάνουν οι χρήστε πολύτιμο χρόνο που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν ε, θεσπίζει τέσσερι καινοτομίε που υποστηρίζω. Υποστηρίζω τη δημιουργία ε, μια νέα ευρωπαϊκή πύλη έρευνα, μέσα στην οποία οι αστυνομικέ αρχέ επιτόπου και οι συνοριοφύλακε μπορούν ταυτόχρονα να εξακριβώσουν όλε τι πληροφορίε μέσω των πληροφοριών που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, αντί να πρέπει να διαβουλεύονται κάθε ε, βάση δεδομένων ξεχωριστά. Και ο εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων είναι κάτι που χαιρετίζω. Έτσι, οι αρχέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω μπορούν να εντοπίζουν την απάτη όσον αφορά τι ταυτότητε. Και χάρη σε αυτό, ε, αυτοί που ε, καταχωρούνται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων διαφορετικό όνομα διαφορετικά θα ξέφευγαν από τον εντοπισμό τους. Χαιρετίζω τη δημιουργία αυτού του κοινού καταλόγου στοιχείων ταυτότητας θα διευκολύνει κατά πολύ τον εντοπισμό των υπηκών τρίτων χωρών ε, που βρίσκονται στην επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, χαιρετίζω τη δημιουργία τη υπηρεσία τη κοινή ε, για την ε, ανταλλαγή βιομετρικών στοιχείων. Να επενθυμίσω ότι κανένα συμπληρωματικό στοιχείο για τους ανθρώπους δεν θα συλλέγεται λόγω διελειτουργικότητας και ότι όλοι οι κανόνες προστασίας των δεδομένων σε κάθε σύστημα θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Κατά κλείδι, θέλω να συγχαρώ τους δύο συνάδελφους για την ποιότητα τη εργασία του και του διαβεβαιώνω ότι θα τύχουν τη υποστήριξη τη ΑΛΔΕ κατά την ψηφοφορία του λόγω κανονισμού. Και κύριε Πρόεδρε, αν αυτό θα έπρεπε τελευταία φορά που παίρνω το λόγο ενώπιον του ημικυκλίου, θα ήμουν ευτυχής να το έχω κάνει μιλώντα πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, κύριε Ντεπχέ. Συνάδελφε Φράντ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για την ε, εγκαθίδρυση της ε, διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών ε, τραπεζών δεδομένων δεν είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Όχι. Έχει υψηλή πολιτική σημασία. Η, ο υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων μας λέει προειδοποιώντα ότι κάνουμε ένα βήμα από το οποίο θα μπορούμε ποτέ να κάνουμε πίσω. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δεδομένων, όταν δημιουργήθηκε η Επιτροπή του άρθρου 29, εξέφρασε τι ανησυχίε γιατί λοιπόν μα προειδοποιούν από αυτό το βήμα οι δικοί μα οι εμπειρογνώμονε, Γιατί η προστασία των δεδομένων ε, βασίζεται στην αρχή του σε τι χρησιμεύει. Δεν χρειάζεται ε, να ανταλλάσσουμε στοιχεία, δεν ξέρουμε σε τι χρησιμεύουν. Αλλά δημιουργούμε τώρα κάτι με αυτόν τον κανονισμό για τη δελτουργικότητα ε, μέσω αυτού του CER που είναι ένα αποθετήριο στοιχείων ταυτότητας όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση διάφορες αρχές. Δηλαδή φτιάχνουμε μια τερατώδη τράπεζα δεδομένων όπου θα έχουμε τα στοιχεία και αθώων συμπολιτών. Συχνά ακούμε το επιχείρημα ότι έχουμε το πρόβλημα της πολλαπλές ταυτότητες. Ε, κυρίως οι συντηρητικοί μας το λένε. Αναφέρουν το παράδειγμα των τρομοκρατών ε, στην αγορά Χριστουγέννων του Βερολίνου. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πούμε κάτι σαφώς. Τον, τον ήξεραν διάφορες υπηρεσίες, τον παρακολουθούσαν. Και αυτό το οποίο πήγε στραβά στο συντονισμό των υπηρεσιών ε, μελετάτε τώρα από μια εξεταστική επιτροπή. Δεν υπήρχε συνδυασμό ε, των ε, ταυτοτήτων του. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα όμω. Και όπως σας είπα, με αυτό το μέτρο δεν θα μπορούμε μετά να κάνουμε πίσω. Αυτό το κεντρικό αποθετήριο θα έχει και τα βιομετρικά. Έτσι όσοι θέλουν να κάνουν hacking θα έχουν ε, με τη μία πάρα πολλά στοιχεία για τα άτομα αυτά και θα μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα. Και ίσως να οδηγήσει αυτό και σε αντιζηλίες μεταξύ των υπηρεσιών. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορώ να εγκρίνω. Διότι στην ουσία θα δημιουργήσουμε μία ε, άσκοπη και ε, ακριβή νέα δομή η οποία Κυρίω θα ωφελήσει αυτού που πουλάνε υπολογιστέ και λογισμικό. Νομίζω ότι πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ το κράτο που θα επιτρεί τα πάντα. Ω πράσινοι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε το πακέτο για την διαλειτουργικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Έρνστ, 1,5 λεπτό. Α θυμηθούμε για άλλη μια φορά την περίπτωση Άμρη. Οι ε, αρχές ασφαλείας απέτυχαν θλιβερά. Όχι επειδή υπήρχε θέμα πολλαπλών ταυτοτήτων διότι η υπηρεσία προστασίας του συντάγματος σταμάτησε να τον παρακολουθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και τι συνέβη. Ότι γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή αρχή για να εντοπίζουμε ταχαίως αυτά τα άτομα. Μα ούτως ή άλλως έχουμε πάρα πολλές ε, τράπεζες δεδομένων. Έχουμε αυτό το, την αντιστοίχηση για τα βιομετρικά στοιχεία του, τον ανοιχνευτή τεχνικών, ε, συγγνώμη, βιομετρικών ε, ε, δεδομένων. Περί τίνος πρόκειται τελικά. Πώς θα περιορίζουμε αυτή την, την τάση των υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα πάντα για τα πάντα. Και όπως είπε και ο προηγούμενος, είμαστε σε ένα σημείο από το οποίο δεν μπορούμε να επιστρέψουμε μετά. Εάν ε, εγκαταλείψουμε μια φορά αυτή την αρχή ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένη η χρήση των στοιχείων, ποτέ δεν μπορούμε να επανέλθουμε. Θα δημιουργήσουμε ένα γενικό κράτος επιτηρητή που θα παρακολουθεί τα πάντα. Και έχουμε και το Eurodac. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η μετανάστευση και η εγκληματικότητα μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Και μήπως θα αξιοποιούμε και τα στοιχεία τρίτων χωρών Στην ουσία τι κάνουμε. Στην ουσία θα ελέγχουμε βιομετρικά τους πάντες. Πρώτα απ' όλα τους υπηκόους ε, τρίτων χωρών, αλλά αύριο και των δικών μας. Καλώς ορίσατε στο θαυμαστό καινούριο κόσμο. Το συνάδελφε Φεράρα, για ένα λεπτό, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πακέτο νομοθετικού περιεχομένου είναι σημαντικότατο. Η δικαστική συνεργασία και η αστυνομική συνεργασία με τη βελτίωση τη ανταλλαγή των πληροφοριών συμβάλλουν στην πράξη στην ενίσχυση, τη σημαντική ενίσχυση τη εσωτερική ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τι τρομοκρατικέ επιθέσει των Παρισίων, ε, περιμέναμε να ζητήσαμε αμέσω παρεμβάσει για να καλύψουμε τα κενά διαχείριση των πληροφοριών και θέλαμε να υπάρχει λειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και να δίνονται πληροφορίε. Η λειτουργικότητα επιτρέπει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των βάσεων δεδομένων θα αντιπροσωπεύσει τώρα πολύτιμη υποστήριξη των εθνικών αρχών του τομέα τη ασφάλεια, των συνόρων και των διαδικασιών, ε, διαδικασιών θεωρήσεων. Θα γίνεται καλύτερη εξεκρίβωση, θα είναι αποτελεσματικότερη έλεγχη στα κράτη-μέλη και έτσι θα διευκολυνθεί ο εντοπισμό εκείνων που αποτελούν απειλή σε αντίθετα με την απάτη της ε, ταυτότητας έρευνα ή δίωξη για σοβαρά δικήματα. Είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί όσο μόνο μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών, αλλά μέσω της καλύτερης διαχείρισης των πληροφοριών ε, και κυκλοφορίας αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ ε, τους εισηγητές Λένς και Κοέλιο για την προσπάθειά τους. Συνάδελφε Νίντερ Μιούλερ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για το έργο τους που βασίστηκε σε εξαιρετική συνεργασία πραγματικά. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Η σοσιαλιστική ομάδα είχε πολλές απόλυτα θεμητές επιφυλάξεις για την μεταρρύθμιση αυτή που κάνουμε όσον αφορά τις βάσεις δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των βάσεων δεδομένων. Είμαι πεπισμένος ότι οι διάφορες ε, βάσεις δεδομένων έχουν δημιουργηθεί για διαφορετικούς σκοπούς και δεν είναι τυχαίο αυτό. Σχεδιάστηκαν έτσι και υπήρχε λόγος που σχεδιάστηκαν έτσι να είναι χωριστές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, δυσκολίε όσον αφορά την ασφάλεια στην Ευρώπη σήμερα και καταλαβαίνω ότι χρειαζόμαστε συστήματα τα οποία θα μα επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τι απάτητε που γίνονται με τι ταυτότητε. Οι αρχέ επίση πρέπει να μπορούν να κάνουν τη δουλειά του καλά. Ναι, αλλά η προστασία τη ιδιωτικότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση των συστημάτων αυτών πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεκτικά. Θέλω επίσης να σας αναφέρω τις επιφυλάξεις τόσο από πλευράς του υπόπτη προσωπικών δεδομένων αλλά και ε, των θεμελιδών δικαιωμάτων όσον αφορά τον εντοπισμό των απατών που γίνονται για τι ταυτότητε. Πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα στου ελέγχου που κάνουμε. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν μπορείτε να υποθέσετε ότι οι τρίτων χωρών είναι μια απειλή για μα εξορισμού. Επίσης ανησυχώ πάρα πολύ για την τάση που έχουμε διαπιστώσει σε σχέση με αυτή την έκθεση όταν μιλάμε για ασφάλεια και κάθε φορά που μιλάμε για ασφάλεια περιορίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εμένα με ανησυχεί αυτή η τάση. Πρέπει να φτιάξουμε μια Ευρώπη όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα και ανησυχίε για την ασφάλεια δεν βρίσκονται σε ανταγωνισμό το ένα με το άλλο, αλλά συνεργάζονται, πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό συμβιβασμό. Στο δύο λεπτά Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι η βάση δεδομένων για μένα ήταν κάτι καινούριο. Όταν ανέλαβα εδώ τα κοντά μου, ήμουν δικηγόρος που ασχολιόμουν με τη μετανάστευση, οπότε πήγαινα συχνά στα σύνορα, ασχολιόμουν με τα θέματα που είχαν να κάνουν με τα σύνορα. Η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση λοιπόν που εγώ θα εξετάσω από τη νομική πλευρά της μετανάστευσης. Πώς βλέπω λοιπόν εγώ αυτή την πρόταση. Είναι το ίδιο όπως η γενική τάση που διαπιστώνουμε τελευταία που εμποδίζει τους ανθρώπους να έρχονται στην Ευρώπη. Αυτού του είδους οι έλεγχοι δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να φεύγει όμως από τις χώρες του. Χρειαζόμαστε να βασιστούμε στις αξίες μας, στις αρχές μας. Αν συνεχίσουμε να υιοθετούμε νομοθεσία που υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν τηρούμε τις αρχές μας. Οι μετανάστες θα συνεχίσουν να έρχονται. Τους φοβόμαστε. Γι' αυτό παραβιάζουμε τα βασικά δικαιώματα για την ιδιωτικότητα. Επίσης, λέμε ότι οι μετανάστες είναι ενδυνάμοι τρομοκράτες, εγκληματίες. Μα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα δικά μου πιστεύω και της ομάδας μου. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα με ανοιχτό μυαλό. Εγώ στην αρχή ήμουν ανοιχτή και ήμουν θετική για την πρόταση, αλλά έτσι όπως τη βλέπω σήμερα αντιβαίνει στις αρχές μου. Το θέμα του αποθετηρίου, για παράδειγμα, ε, δεδομένων ταυτότητας ή η υπηρεσία της τύχησης βιομετρικών δεδομένων. Είναι μια κεντρική βάση δεδομένων που θα εξυπηρετεί όλε τι υπόλοιπε. Μα πάει πολύ μακριά αυτή η υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάει πάρα πολύ μακριά και δεν μα πείθει ότι πραγματικά χρειάζονται όλα αυτά, ότι είναι αναγκαία, ότι είναι αναλογικά. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα επειδή έχουμε ένα στόχο. Πρέπει να βασιστούμε στις αρχές μας και στις αξίες μας και συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε πριν ότι πρόκειται για μια τερατώδη βάση δεδομένων. Πιμέντα Λόπες τώρα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει να συλλέξουμε βιομετρικά στοιχεία και άλλα και θα υπάρχει ανταλλαγή προφοριών και εναρμόνιση του τρόπου συλλογής τους για να είναι πιο εύκολο οι αρχές να τις ανταλλάσσουν χωρίς ε, να χρειάζεται η άδεια ενός δικαστή. Δεν είναι τεχνικό θέμα, είναι ουσιώδης πολιτική πράξη που δημιουργεί ένα σύστημα πλήρους επιτήρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα την ελευθερία των πολιτών. Και δημιουργεί μια σύγχυση των σχέσεων μεταξύ μετανάστευσης, τρομοκρατίας, εγκληματικότητας. Στην ουσία υπάρχει ε, υπόθεση ενοχής. Οποιοδήποτε θεωρείται ε, ενδεχόμενα εγκληματίας. Τώρα οι πολίτες τρίτων χωρών και ε, αύριο και οι δικοί μας πολίτες. Είναι απαράδεκτη αυτή η ξενοφοβική και ρατσιστική αντίδραση στην ε, μετανάστευση. Όλα αυτά είναι ένα παράδειγμα που δείχνουν ότι η ακροδεξιά έχει βρει γόνιμο έδαφος. Η κυρία James η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στοχεύει στον έλεγχο. Και τι καλύτερο μηχανισμό και τι το τελευταίο παράδειγμα από το τελευταίο παράδειγμα που χωνοποιών μα. Μαζί με άλλου συναδέλφου που ήδη μίλησαν, εγώ θεωρώ ότι αυτή η προέγγιση είναι και λανθασμένη και έχει λάθο στόχο. Και χειρότερα είναι και αναποτελεσματική από πλευρά κόστου. Το κόστο αυτή τη νομοθεσία για τον φορολογόμενο τη Ένωση είναι 460 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνεται το αυτό με αυτά που δαπανούν οι ΗΠΑ ε, που έχουν ένα παρόμοιο πληθυσμό για να προστατεύει την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών της. Είναι στάγονο στον ωκεανό. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει σοβαρά να προστατεύσει τους πολίτες της, τότε χρειάζεται ένα σοβαρός και αναλυτικός και στοιχειοθετημένος προπολογισμό. Άλλοι είπατε μια άλλη ανησυχία. Η ποιότητα των στοιχείων για να έχουμε μια ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για να ε, συγκεντρώνουμε και να συγκεντρωνοποιούμε να υπάρχει συγκεντρωτική ε, χρήση των βιομετρικών στοιχείων έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα των στοιχείων που θα συλλέγουμε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ότι οι εγκληματίες καταστρέφουν τις ταυτότητές τους, δεν υπάρχει καμία ενεχνευσιμότητα της ε, δράσης τους και άρα δεν μπορούμε να τους συλλάβουμε. Τα ευρωπαϊκά διαβατήρα, όπως ξέρετε, πουλούνται στη μαύρη αγορά. Και υπάρχουν ε, μεγάλοι αριθμοί τέτοιων διαθέσιμων. Και κανείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συζητήσει σε επίπεδο ε, Συμβουλίου επίσης πώς δυνατόν 500 πολίτες της Ένωσης να αισθάνονται καλά για το ότι συλλέγονται τα στοιχεία τους, τα διαχειρίζονται και έχει κανείς πρόσβαση σε αυτά. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην θέλει να γίνει αστυνομικό κράτος. Αλλά πρέπει να το θέσω ως ερώτημα. Μήπως το θέλει. Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι ο πυλώνας, ε, ο τόσο σημαντικός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απειλείται. Αυτή η νομοθεσία είναι απλώς περισσότερος έλεγχος. Θα αρκούσε ο έλεγχος από κυρία Χακράτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τζέμς. Μωρά, ένα λεπτό. Οπότε ο συνάδελφος Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Κίνγκ, κύριε Επίτροπε Βραμόπουλε. Ως Ισπανός Σοσιαλιστής και Ευρωπαίος στηρίζω οποιαδήποτε ρύθμιση η οποία ε, διασφαλίζει προστασία από την εγκληματικότητα, από την τρομοκρατία, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες των πληροφοριών. Τι είναι η διαλειτουργικότητα βοηθάει όλες οι βάσεις δεδομένων να διασυνδεθούν όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Είτε πρόκειται για ε, τις θεωρήσεις, είτε πρόκειται για το Eurodac, το Schengen, αλλά και όλες τις τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με το αίτιας, με τις εισόδους-εξόδους και το τέκρις επίσης. Όμως, εγώ θέλω να τονίσω το θέμα των εγγύσεων. Θα πρέπει να προσέξουμε τα εξή. Πρώτον, να μην μπερδεύουμε τη μετανάστευση και την τρομοκρατική απειλή. Δεν είναι το ίδιο. Δεύτερον, να τηρούμε πλήρως τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που μιλάει για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Τρίτον, να τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα για το ΚΑΤΣΤΙΑΕ, οπότε τώρα ο Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους που έλαβαν το λόγο για τον ενδιαφέρον και την προσπάθεια που καταβάλλετε για αυτά τα θέματα.